κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίσω την έναρξη των ε, εργασιών μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ε, ιού του AIDS από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι μετά από τη δήλωση της Επιτροπής θα ακολουθήσει ένας γύρος ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και ότι δεν θα διεξαχθεί διαδικασία Catch the Eye. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ντάλι εξ ονόματος της Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι σήμερα. Sorry. Σήμερα το βράδυ υπομιλητής ε, πρόκειται για λαθάκι. Στην Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για το